όταν Αν χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο τα δεδομένα, καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει η δυνατότητα για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα να μην ισχύει. Η πρόταση της Επιτροπής είναι μια ποσοτική προσέγγιση και όχι ποιοτική προσέγγιση. Μιλάει για μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οργανισμοί έχουν κάπου 250 υπαλλήλους, λέει, και έχουν πιο αυστηρούς κανόνες. Εμείς πιστεύουμε ότι ανταυτού θα πρέπει τα τετριμένα δεδομένα και τα ευαίσθητα δεδομένα να τυχαίνουν διαφορετικής προσέγγισης από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο κανονισμός θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη δεδομένων τα οποία απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις όπου η χρήση των προσωπικών δεδομένων δεν αφορά πάντα ευαίσθητα δεδομένα. Στο μέλλον λοιπόν χρειάζεται ένας χώρος απλοποιημένων κανόνων για την καθημερινή ζωή, για τα τετριμένα δεδομένα και όχι για τα ευαίσθητα δεδομένα. Η μεταρρύθμιση της οδηγίας κατά τη γνώμη μας ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτή την ανάγκη. Το Συνδικό Κοινοβούλιο συνεπώς προτιμάει ελεύθερη χρήση δεδομένων εφόσον δεν παραβιάζεται η ακαιρότητα του ατόμου. Ένας κανονισμός σαν αυτόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί και σε περισσότερη γραφειοκρατία, σε πιο λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερο κόστος για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν είναι ευαίσθητα. Μία προσέγγιση μονοθυρική δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Η πρόταση της Επιτροπής επίσης όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης σε πολλούς τομείς, πάρα πολλούς ε, τομείς από ό,τι βλέπουμε τώρα, είναι επίσης πρόβλημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που κάνει είναι ότι κάνει μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση του νομοθέτη, αν θέλει ίδια να γίνει νομοθέτης. Αυτό αντιβαίνει στη συνθήκη. Έπειτα ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο κανονισμός στο μέλλον. Κάτι το οποίο αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Η ποσότητα των κατεξουσιοδότηση πράξεων, κατά τη γνώμη μας, είναι υπερβολικά μεγάλη. Και στην πράξη οι εθνικές αρχές χάνουν μέρος της ανεξαρτησίας τους. Γιατί τελικά πρέπει να λαμβάνουν εντολή και διαταγές εντό αγωγικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο στη Σουηδία θα αποτελέσει συνταγματικό ζήτημα. Και φαντάζομαι όχι μόνο στη Σουηδία και σε άλλε χώρε. Ένα κατακλείδη. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπω προτείνεται, είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό, με υπερβολικέ λεπτομέρειε και θα οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα και περιτές δαπάνες. Αλλά πιο σημαντικό δεν θα έχουμε την καλή προστασία δεδομένων που πραγματικά χρειάζεται. Χάνει την ευκαιρία έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια σύγχρονη και αποτελεσματική πρόταση. Χάνεται σε λεπτομερείς ρυθμίσεις. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι πολίτες να δεχτούν την προτινόμενη μέθοδο. Παρόλο που ο κόσμος πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη προστασία των δεδομένων. Επιτρέψτε μου να σας πω και δύο λόγια όσον αφορά την εποπτεία. Γιατί μας ρωτάτε και για τις εποπτικές αρχές. Η Σουηδική Αρχή Εποπτείας Δεδομένων έχει ικανοποιητικούς πόρους. 5 εκατομμύρια ευρώ για του χρόνου, για παράδειγμα, στον προπολογισμό προβλέπονται αλλά εννοείται ότι οι ανάγκες βαίνουν αυξανόμενες και πολύ πιθανό να χρειαστούν περισσότερα χρήματα ακόμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Έριξον. Ο κύριος Χάστινγκς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία μου. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πακέτο που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα μπρος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι ευπρόσδεκτο. Συγχρόνως όμως έχει και πολλές αδυναμίες. Πρώτα απ' όλα το πακέτο αυτό δεν είναι τόσο πλήρες όσο θα έπρεπε να είναι. Και έπειτα, τόσο αναφέρονται για την επιβολή του νόμου δεν αποτελούν επαρκή προστασία. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία θα έπρεπε να διευκρινιστούν περισσότερο. Εμείς έχουμε αναπτύξει την τοποθέτησή μας βάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και χαίρομαι που πολλές από τις παρατηρήσεις μας έχουν συμπεριληφθεί και στο κείμενο του εισηγητή και τα είπανε και πολλοί χτες. Δεν θα τα επαναλάβω. Σήμερα μιλάμε για μια αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος και των υποχρεώσεων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα καταχωρημένα άτομα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ε, ασκούν τα δικαιώματά τους στην πράξη και να έχουν και τις ε, πηγές που χρειάζονται και από την άλλη μεριά και τις υποχρεώσεις τους θα πρέπει να μπορούν όλοι να τις φέρουν σε πέρας. Άρα και οι δύο αυτές πλευρές θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Εξού και μιλάμε για την εποπτεία και την επιβολή και συγχρόνως μιλάμε και για την συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ αρχών προστασίας ε, δεδομένων. Γι' αυτό και θα σας αναφέρω από αυτόν 6-7 ε, σημεία. Πρώτα απ' όλα, στηρίζω έντονα τις ε, διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ανεξαρτησία, με την, τις εξουσίες και τους κατάλληλους πόρους που πρέπει να έχουν οι αρχές προστασίας δεδομένων. Είναι κάτι πολύ βασικό για να υπάρχει πραγματικά αυτή η προστασία δεδομένων όπως αναφέρεται στη χάρτα και αυτό το έχει υπογραμμίσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ε, υπόθεση ε, με την Γερμανία, Επιτροπή Γερμανία. Τώρα, με ποιο τρόπο ορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου. Αυτό γίνεται είτε από τις κυβερνήσεις είτε από το Κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν προτιμότερο να προβλέπεται η συστηματική ανάμιξη των εθνικών κοινοβουλίων στον ορισμό των ε, μελών. Όσον αφορά τώρα τους κατάλληλους πόρους, εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν κάπως πιο αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι επαρκούν. Αλλιώς στην πράξη υπάρχει ο κίνδυνος οι πόροι να μην επαρκούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις λεπτομέρειες, υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός για να εμφυσίσουμε περισσότερη αντικειμενικότητα στις ρυθμίσεις. Έρχομαι τώρα στις, κυρίσεις, στις κυρώσεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη ελαστικότητα στις διοικητικές κυρώσεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αναλογικότητα των προστήμων αυτών καθ' αλλά συγχρόνως να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και οι άλλες ε, εξουσίες, οι οποίες μπορεί να μην αναφέρονται ρητά, αλλά σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα διαφορετικών ε, εργαλείων. Σίγουρα να υπάρχει η συμμόρφωση, αλλά όχι μόνο. Χρειάζεται να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά. Το Συμβούλιο πάντως το Ευρωπαϊκό Προστασίας Δεδομένων να ξέρετε ότι θα το κάνει και θα φροντίσει να προτείνει περισσότερη ελαστικότητα αντί να επιβάλλονται κάθε φορά πρόστιμα και μόνο. Τώρα τόσο αναφέρονται για τις ε, αρχές των χωρών μελών. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε λιγάκι τον ορισμό της κύριας εγκατάστασης. δεν ισχύει πάντα το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Μερικές φορές μπορεί να υπάρχει μια κύρια εγκατάσταση σε μια περιοχή της Ευρώπης και όχι σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Τι σημαίνει το lead authority και ποιος είναι ο ρόλος και κατά πόσο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ηγετική αρχή στο θέμα της προστασίας των δεδομένων, να υπάρχει συνεργασία με άλλες ε, αρχές. Δείτε και το κεφάλαιο 7 που μιλάει για τη συνεργασία και τη συνοχή. Η ηγετική αυτή αρχή μπορεί να είναι ηγετική, αλλά μπορεί να μην έχει τις εξουσίες να ασκήσει εκτός της δικιάς της δικαιοδοσίας τις εξουσίες της αυτές. Είτε πρόκειται για επιθερήσεις είτε πρόκειται για την επιβολή του νόμου. Άρα χρειάζεται συνεργασία με άλλες αρχέ. Και ίσως θα ήταν καλύτερο η, η ηγετική αυτή αρχή να συνεργάζεται με άλλες. Τώρα έρχομαι γενικότερα στο κεφάλαιο 7. Νομίζω ότι έχει μια καλή δομή. Υπάρχουν όμως μερικά σημαντικά στοιχεία εδώ που θα ήθελα να διευκρινιστούν και να διορθωθούν ίσως. Έρχομαι τώρα στον μηχανισμό συνοχή συμβατότητα. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπαίνει σε λειτουργία ο μηχανισμός αυτός. Ποιε προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν. Αν σκεφτείτε τις συνέπειες, υπάρχει ο κίνδυνος ο μηχανισμός αυτός να φορτωθεί υπερβολικά. Ή υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει μία κύρια υπόθεση και να υπάρχουν μετά και διάφορες υποϋποθέσεις και να καταλήξουμε σε μεγάλη γραφειοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη ελαστικότητα κάθε φορά που μιλάμε για την υιοθέτηση των ε, αποφάσεων του Συμβουλίου. Ε, θα είναι δύσκολο σε ένα μήνα να καταλήξουμε σε συνένεση ακόμα και για τις καλύτερες ε, δυνατόν σκέψεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε εδώ πιο ελαστικοί και ευέλικτοι. Έρχομαι τώρα στις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφερθήκαμε σε αυτές γενικά χτες. Σε αυτό το μηχανισμό οι εξουσίε τη Κομισιόν πρέπει να είναι περιορισμένε και διευκρινισμένε. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σημαντικό αλλά να περιορίζεται είτε το να υποβάλει στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μια υπόθεση, να έχει και την αρμοδιότητα να υποβάλει γνωμοδοτήσεις. Αλλά άπαξ και το Συμβούλιο έχει αποφασίσει κάτι, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ανατρέψει τις αποφάσεις που παίρνει σε διάφορες υποθέσεις στο Συμβούλιο. Ενώ τώρα αυτό γίνεται και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε και παραβιάζει επιπλέον πιστεύω την αρχή της ανεξαρτησίας έτσι όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Κομισιόν Γερμανία. Συνεπώς, στη συνθήκη αναφέρεται ότι και η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη. Φυσικά και είναι ανεξάρτητη απέναντι στα κράτη-μέλη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει παραβίαση. Έπειτα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου πρέπει να αναμειχθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είτε στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιπροσφυγή, αν κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, είτε να ζητήσει προσωρινά μέτρα. Μια παύση για παράδειγμα. Χτες η κυρία Ρέντινγκ αναφέρθηκε σε προφανείς περιπτώσεις παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου. Ποια είναι η επιχειρηματολογία των ε, εθνικών κυβερνήσεων της Γερμανίας, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ δεν θα στοιχημάτιζα πάντως. Η γραμματεία τώρα του Συμβουλίου ε, Προστασίας Δεδομένων πρέπει να πάρει σάρκα και οστά. Θα μπορούσαμε να παίξουμε αυτό τον ε, ρόλο εφόσον υπάρχουν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που χρειάζονται. Σήμερα η εκτίμηση είναι περιορισμένη. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Να υπάρχουν επαρκείς πόροι. Μπορεί να μην είναι θέμα νομοθεσίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό για να πετύχει η πρόταση. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά εγώ θα αφήσω τον Γιακοπ Κόνστα να μιλήσει γι' αυτό. Μια που έχει εγκρίνει η ομάδα 29 πρόσφατα μια γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνατε την ευκαιρία να μιλήσω Ολλανδικά, να που μπορώ. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, εδώ συγκεκριμένα, είναι αυτό και με το οποίο θα ασχοληθώ εγώ, λέει ο κύριος ε, Κόνσταμ. Είμαστε η ομάδα 29 και έχουμε μία γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία γνωμοδότηση που μάλιστα την βρίσκεται και εδώ, στο τραπέζι, στην είσοδο της αίθουσας. Στην γνωμοδότηση αυτή υπάρχουν και πράγματα βέβαια που δεν έχουν να κάνουν άμεσα με το θέμα που συζητάμε τώρα, αλλά το βέβαιο είναι ότι έχουν μεγάλη σχέση με την ε, προστασία δεδομένων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του ορισμού των ε, δεδομένων, κάτι που συζητήθηκε χτες, ή έχει να κάνει με την ε, απέτηση της ρητής άδειας, το οποίο συμπεριλαμβάνουμε στην ε, γνωμοδότησή μας, γιατί έχει τεθεί πολλές φορές στις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, θα έρθω και στο κατεξοχήν θέμα που μας απασχολεί τώρα και που απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η νέα νομοθετική πρόταση και πόσο πλήρης είναι αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει δύο μέσα, κανονισμό ή οδηγία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εξεταστεί το θέμα ως πακέτο και να δούμε και τις δύο περιπτώσεις. Αρκεί να υπάρχουν οι ίδιες εγγύσεις και η ίδια προστασία. Πρώτο που θέμα, κυρώσεις. Από πλευράς του επόπτη και της επεξεργασίας του επόπτη, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα που πολύ φτηνά αποκτώνται, το είπε και η κυρία Ρέντινγκ. Από το Facebook, για παράδειγμα. Επίσης, πολύ συχνά, εμπορικές επιχειρήσεις ορισμένες χώρες μέλη προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα και καταλαμβάνουν ένα τέτοιο μεγάλο μέρος της αγοράς που καταλήγουν σε μονοπόλιο. Τέτοιες πρακτικές μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το θέμα των ε, κυρώσεων είναι κάτι που πρέπει να το δούμε εντελώς ε, διαφορετικά, όπως είπε και ο κύριος Σούστινγκ. Το θέμα τώρα του μηχανισμού συμβατότητας, συνοχής. Βέβαια, ο κύριος Χούστινγκ τα είπε πάρα πολύ καλά πριν από μένα, αλλά θέλω και εγώ να προσθέσω εδώ δύο σημεία. Πρώτον, δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι για να ξεκινήσει ο μηχανισμός αυτός μεταξύ των διαφόρων ε, εθνικών αρχών περνάει αρκετός καιρός. Ελπίζουμε πάντως σύντομα να έχουμε μία γνωμοδότηση συγκεκριμένη για αυτό το θέμα. και κάτι άλλο για τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναμειγνύεται. Δεν ε, συμφωνούμε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ότι πρόκειται για παραβίαση της ανεξαρτησίας. Έρχομαι τώρα στο θέμα του προπολογισμού. Μίλησε και σου Σουηδό ο συνάδελφος ε, πριν γι' αυτό. Για να υπάρχει αποτελεσματική προστασία, το θέμα αυτό του προπολογισμού αποτελεί τον αδύναμο κρίκο. Και μπορεί με τον μηχανισμό συνοχής πολύ σύντομα να αποτελέσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα διότι όλο και περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται, είναι περιττό να το πω αυτό, ότι την τελευταία δεκαετία έχουν συγκεντρωθεί φοβερά πολλά δεδομένα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για να υπάρχει εποπτεία και να γίνεται η σωστή επεξεργασία αυτών, εννοείται ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα και εναρμόνιση της νομοθεσίας. Αν λοιπόν δεχόμαστε ότι χρειάζεται η εναρμόνιση αυτή, ο μηχανισμός αυτός σημαίνει ότι κάθε αρχή εποπτική πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και άρα η ομάδα εργασίας 29 θέλει να υπάρχει ένα σαφέστερο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο εύρος και περισσότερη ανεξαρτησία από το ΑΕΠ, από την κύρια εγκατάσταση κτλ. Θέλουμε φυσικά ισορροπία στον προπολογισμό του Συμβουλίου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες εθνικές υπηρεσίες οι οποίοι είναι συνήθις ε, ύποπτοι και να δούμε τι έχει γίνει με τον δικό τους προπολογισμό. Τώρα έρχομαι στις κατεξουσιοδότηση ή εφαρμοστικές ε, πράξεις. Συμφωνώ ότι υπάρχει περιθώριο για παρετέρω βελτίωση. Άρα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια για να δούμε πώς θα χρησιμοποιούνται κατά εξουσιοδότηση πράξεις. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να δούμε